Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε τώρα νομίζω να ξεκινήσουμε την κοινή μας συνεδρίαση μαζί με την Επιτροπή Επασχόλησης, όπως γνωρίζετε, αυτό, αυτή προβλέπεται από τον κανονισμό του Six την έναρξη του νέου εξαμήνου, και από τον οικονομικό διάλογο με την Κομισιόν για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης και την ε, έκθεση του μηχανισμού ειδοποίησης. Έχουμε και ένα ολόκληρο πακέτο δηλαδή, έχουμε και τις συστάσεις και είναι πάρα πολύ θετικό που μπορούμε να προβούμε σήμερα σε ανταλλαγή απόψεων μαζί με την διαπραγματευτική μας ομάδα, τον εισηγητή μας, τους εισηγητές μας, συγγνώμη, που θα μπορέσουν να ξεκινήσουν την εκμόνηση της έκθεσής τους. Να καλωσορίσω λοιπόν τον Αντιπρόεδρο τον Πρόσκη, την Επίτροπο Τάισεν και τον Επίτροπο Μοσκοβισή. Όπως γνωρίζετε, η ετήσια έκθεση ανάπτυξης δείχνει μια μετριοπαθή ανάπτυξη ανάπτυξη, ανάκαμψη, διατηρεί τις ε, κεντρικές προτεραιότητες ε, της πεσινές επενδύσεις, διαστοτικές μεταρρυθμίσεις, ε, δημοσιονομική εξυγίανση και φυσικά τώρα πώς θα, θα εφαρμοστούν αυτές οι προτεραιότητες συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό κύκλο είναι ένα σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα. Και ξέρετε ότι έχουμε το πρώτο βήμα για την εξηγήνση καθώς και με τον ε, μηχανισμό άγγελης προειδοποίησης καθώς και με τη διαδικασία ε, ισορροπίας όπου τα δύο στοιχεία συνδυάζονται μεταξύ τους και θα αρχίσουμε με τις εισηγήσεις των τριών επιτρόπων και θα συνεχίσουμε με ερωταπαντήσεις. Αλλά πριν από αυτά, Μαρίσα, θες να προσθέσεις κάτι. Ευχαριστώ κύριε Γκολτιέρη. Καλώς ορίσατε επίτροποι, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι. Αρχίζουμε με αυτή την κοινή περιπέτεια πριν από κάνα χρόνο, όταν συζητήσαμε την οικονομία, αλλά όχι μόνο την οικονομία, τη συζητήσαμε μέσα στο πλαίσιο της απασχόλησης, διότι αν έχουμε 23 εκατομμύρια ακόμα ανέργους εντός της Ένωσης ξέρεις σαφώς ότι αυτό πρέπει να το καταπολεμήσεις και η οικονομία είναι το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το κοινό στόχο της κοινωνικής Ευρώπης. Και γι' αυτό και ε, αυτή η συνεργασία είναι τόσο πολύ σημαντική για μας, γιατί αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, είναι πιο εύκολο να επιτύχουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε σήμερα εδώ και προσβλέπω στις ερωτήσεις αλλά και κυρίως στις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά αυτά που είπε. Κοινό μα στόχο είναι το να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη και τι θέσει απασχόληση. Και βεβαίω ε, αυτά που μπορούμε να διαβάσουμε στην έκθεση του μηχανισμού προειδοποίηση, αυτή η έλλειψη ισορροπία ανάμεσα στην πρόσβαση ε, ε, στι χώρε επενδύσει και τι και τις δημόσιες αποταμιεύσεις μάλλον και τι επενδύσει, είναι ενδεικτική. Σας ευχαριστώ κύριε Σοντομπρόφσκη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πακέτο στις 26 Νοεμβρίου, το φθινοπορεινό, σηματοδοτώντας όπως συνήθως και την άρξη του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το πακέτο για φέτος περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία στο εξάμεινο, τα οποία την, στην ανακοίνωσή μα στις 21 Οκτωβρίου την ολοκλήρωση της οικονομικής και Νοσματικής Ένωση τάση και αγραφήσαμε. Επρόκειτο για μια ανακοίνωση που αφορούσε την εφαρμογή της έκθεσης των πέντε προέδρων. Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης και των βελτιώσεων. Για πρώτη φορά φέτος είχαμε μία ε, συζήτηση στην Ολομέλεια στις 11 Νοεμβρίου, εδώ στο Κοινοβούλιο, πριν από τη δημοσιοποίηση του πακέτου. Η συζήτηση μας έδωσε σημαντικά σχόλια ε, και σημαντική ήταν η συνεισφορά του. Λάβαμε λοιπόν όλα τα σχετικά σχόλια υπόψη μας ε, στην οριστική έκδοση του εγγράφου μας. Και πάνω σε αυτό ε, θα βασιστούμε για να έχουμε μεγαλύτερη νομιμοποίηση, λογοδοσία και οικειοποίηση, διοκτησία. Να έρθω στην ουσία του πακέτου που υποβάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το πακέτο αυτό λοιπόν αποτελείται από την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη το 2016, για τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της πολιτικής μας για τον επόμενο χρόνο. Έχουμε και το μηχανισμό επαγρύπνησης. Ε, πρώτη φορά έχουμε αυτή την έκθεση για την, ε, τον εντοπισμό πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών, την κοινή έκθεση για την απασχόληση που αναλύει την κατάσταση της απασχόλησης στα κράτη-μέλη και ποιε είναι οι απαντήσει που δίνουν τα κράτη-μέλη με τι πολιτικέ του και έχουμε και τις συστάσει για την Ευρωζώνη που φέτος ε, νωρίτερα δημοσιοποιήθηκαν τον Νοέμβριο για να δείξουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση και ανάγκη σύγκλησης μεταξύ των χώρων της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η καινοτομία της ε, φετινής χρονιάς, ότι οι συστάσεις για την Ευρωζώνη υποβάλλονται ήδη από φέτος, ήδη από τώρα, για να μπορούν τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους ε, όταν συντάσσουν τα ειδικά αναχώρα έγγραφα να λαμβάνουν λοιπόν τις συστάσεις αυτές υπόψη και για να δούμε έπειτα και ποιες είναι οι κοινέ προκλήσεις ε, στις χώρες της Ευρωζώνης ε, για να υποδοθούν και οι συστάσεις σχετικές ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης με βάση τις παρατηρήσεις μας. Για το 2016 τώρα την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητε πολιτικές που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη και να ενισχύσουν και τη σύγκληση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις χαμηλές τιμές ε, των βασικών αγαθών ε, και να ε, αξιοποιήσουμε τις χαμηλές αυτές τιμές και να ενισχύσουμε και τις άλλες πολιτικές μας για να έχουμε βιωσιμότητα. Θεωρούμε ότι οι οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες το 2015 της σχετικής επισκόπησης για την ανάπτυξη παραμένουν εγκαιρές στο μεγαλύτερο μέρος τους. Το 2016 λοιπόν ουσιαστικά συνεχίζουμε με βάση τις ίδιες προτεραιότητες οι οποίες είναι να έχουμε περισσότερη όθηση στις επενδύσεις, μεταφορι... ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επίφθηνες, υπεύθυνες φορολογικές πολιτικές. Και θέλουμε επίσης ε, τα οικονομικά και κοινωνικά επίπεδα να προσεγγίσουν το ένα το άλλο και να πλησιάσουν τους στόχους μας για τις ε, μέγιστες δυνατές επιδόσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ε, το σχέδιο για τις επενδύσεις στην Ευρώπη μπαίνει σε τροχιά και μετά τη δουλειά του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα εμπόδια για τις επενδύσεις. Θέλουμε να τονώσουμε τις δημόσιες ε, και ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση για να ενισχύσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Και πέραν αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα ένα σημαντικό βήμα με την πρότασή τη ε, για έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εγγύηση Καταθέσεων και για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων ε, στον τραπεζικό τομέα. Εστιάζουμε στην ε, δημιουργία θεμελίων για την ανάπτυξη και την θέσει εργασία. Άρα πρέπει να εφαρμόσουμε τις σωστές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μιλάω και για την αγορά προϊόντων και για την αγορά εργασίας, για τη δημόσια διοίκηση. Πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την καινοτομία. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που εντάσσονται και στην ευρύτερη προσπάθεια πολλών κρατών μελών για να διορθώσουν τις ανισορροπίες και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε τομείς σημαντικούς για την παραγωγικότητα και τη σύγκληση. Έχουμε το μηχανισμό επαγρύπνηση του 2016. Δείχνει αυτό ο μηχανισμό ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη τη μακροοικονομικέ ανισορροπίε που εντοπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, παραμένουν ε, κάποιοι τομεί ανησυχία. Ε, Παραδείγματο χάρη, υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέο σε πολλά κράτη-μέλη που αποτελεί και μια πηγή ευαλωτότητα και καθυστερεί την ανάπτυξη σε κάποιες χώρε μάλιστα ανακύπτουν και νέες προκλήσεις. Ε, στο πακέτο δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ε, στα θέματα της ε, απασχόληση και στα κοινωνικά ζητήματα. Θα πρέπει να έχουμε και ευελιξία, αλλά να παρέχουμε και ασφάλεια ταυτόχρονα, να βρούμε δηλαδή την σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο. Η κρίση έδειξε ότι έχει διαβρωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτέ είναι βασικέ αξίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία αποτελούν προποθέσει για την αποκατάσταση κοινωνική δικαιοσύνη. Τώρα, το σχέδιο τη κοινή έκθεση για την απασχόληση δίνει περισσότερε πληροφορίε ε, σε σχέση με του στόχου αυτού. Τρίτο πυλώνα πολιτική τη ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη. Υπεύθυνε φορολογικέ πολιτικέ. Έχουμε το μέσο έλλειμμα, ε, το δημοσιονομικό στην Ευρωζώνη που συνεχίζει να μειώνεται. Αναμένεται να ανέρχεται στο 1,7% το ΕΠΑ για του χρόνου. Και το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη και αυτό αρχίζει να μειώνεται από φέτος. Όμως είναι σημαντικό να έχουμε δημόσια, ε, συγγνώμη, βιώσιμα δημόσια οικονομικά και να αφήσουμε και κάποιο φορολογικό χώρο διαθέσιμο εκεί που είναι αυτό δυνατό. Θα πρέπει να δεθούν κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων εργασία, να είναι δίκαιο το φορολογικό σύστημα. Θέλουμε επίση και ένα εξυγχρονισμένο σύστημα κοινωνική ασφάλιση που θα ανταποκρίνεται στι προκλήσει ενό γυράσκοντο πληθυσμού. Χρειάζεται λοιπόν δράση κατεπηγόντω στου τομεί αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επειδή υπάρχει ε, αλληλεξάρτηση και ίσως εκείνο επιμόλυνση από το ένα κράτος ε, μέλος στο άλλο θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός των οικονομικών πολιτικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά τώρα τις συστάσεις για την Ευρωζώνη. Εκεί εστιάζουμε σε σημαντικά ζητήματα για μια εύρυθμη ε, Ευρωζώνη και προβλέπουμε και συγκεκριμένες συστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ε, προσαρμοστικότητα, σύγκληση, μέτρα που έχουν να κάνουν με το ε, υψηλό χρέος το οποίο κληρονομήσαμε από, τη χρήση, από την κρίση. Θέλουμε επίσης ένα υγιές εύρο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε και την Οικονομική και Νοσματική Ένωση. Η παγίως της ανάπτυξης ε, ε, θα πετύχει αν όλα τα θεσμικά όργανα και όλα τα κράτη-μέλη συνεργαστούν. Βέβαια αυτό ε, απαιτεί και την στενή συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, εθνικών περιφερειακών τοπικών αρχών, εθνικών κοινοβουλίων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κοινωνίας των πολιτών. Προσβλέπω στη στενή αυτή συνεργασία για τα ζητήματα που σας προανέφερα και προσβλέπω και στη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας είπατε και για το σύστημα αυτό SA το οποίο ε, συνεχεί άρχισε να δρομολογείται γιατί δεν είχαμε κάποια ε, μάλλον για το ΕΦΣΙ συγγνώμη μας είπατε το ΕΦΣΙ αρχίζει να δρομολογείται και αυτό είναι σημαντικό δεν είχαμε στοιχεία ο Πιέρ Μασκοβισή είναι επόμενος ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για αυτή τη νέα εκδοχή του οικονομικού διαλόγου. Είχαμε εξάλλου μιλήσει για την έγκαιρη, για, για τον μηχανισμό προειδοποίησης που χαίρομαι να σας παρουσιάσω και να εστιαστώ στα όσα είναι νέα σε σύγκριση με τα όσα έγιναν το περασμένο χρόνο και όσον αφορά την παρακολούθηση του, τη συνέχεια που θα δοθεί το 2016. Πρόκειται για τον, την ανάλυση του κύκλου των ανισορροπιών της περασμένης χρονιάς, τα κράτη, να εντοπίζει τα κράτη-μέλη που μπορεί να επηρεαστούν από αυτή την έλλειψη ισορροπίας, και, αλλά πρόκειται για μόνο μία εκκίνηση. Πρέπει να γίνει η βάθος ανάλυση και μετά η Κομισιόν καταλήγει στην ύπαρξη ή όχι της υπερβολική ή όχι ε, ανισορροπία. Σήμερα προσέχουμε ιδιαίτερα ε, της, ε, τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. Τονίζουμε την αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα στις οικονομίες της Ευρωζώνης και δύο συμπεράσματα θα πρέπει εδώ να τονιστούν. Καταρχήν υπάρχει πλεόνασμα στον τρέχοντα λογαριασμό της Ευρωζώνης που είναι ένα από τα πιο σημαντικά στον κόσμο και αυτό δικατοπτρίζει κυρίως οι υπερβολικές εγχώριες αποταμιεύσεις σε σύγκριση με τις επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, η πίεση που ασκείται για τη μείωση του χρέους εξακολουθεί να πιέζει την ανάκαμψη. Αυτό είναι αλήθεια για τις χώρες που είναι χρεωμένες, αλλά και για αυτές που είναι λιγότερο χρεωμένες. Και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάκαμψη. Η Μαρία θα μας μιλήσει τώρα και για την ενίσχυση της κοινωνικής πτυχής. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν έρθει σε διαβουλέ στη τεχνική προπαρασκευή και έχουν προσθεθεί τρεις ε, ε, παρατηρήσεις που σχετίζονται με την απασχόληση. Αυτό η καινοτομία δεν αφαιρεί την εστιασμό από τις ε, διαδικασίες επίγουσας ανάγκης. Προσπαθούμε να κάνουμε τις διορθώσεις, να βλέπουμε τις νέους δείκτες, αλλά αυτοί δεν σημαίνουν από μόνοι τους την αναθεώρηση της μικρομεσαίας ε, ε, κατάστασης. Έχουμε επιλέξει 18 κρατημέλη για εις βάθος ανάλυση, τα 16 θα ε, υποβληθούν στην ε, αναθεώρηση του χρέους γιατί φάνηκε ότι είχαν υπερβολικές ανισορροπίες σε πέρυσι. Επίσης, η βάθος ε, μελέτη θα γίνει για πρώτη φορά για την Αυστρία και την Εστονία. Όσοι ήθιστε αυτές οι αποφάσεις για το κατά πόσο οι ανισορροπίες ή οι υπερβολικές ανισορροπίες υπάρχουν θα το δούμε στην Κομισιόν όταν θα δημοσιεύσουμε την εις ανάλυση το Φεβρουάριο. Τώρα, όπως και εσείς τονίσατε, ε, επανειλημμένα θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή και θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ευρωπαϊκή διάσταση, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Έχουμε ε, πολλές συστάσεις ε, για το εξάμεινο μαζί με το IGS, δηλαδή πολύ πριν από τις αναχώρα συστάσεις. Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει καλύτερη ένταξη των εθνικών διαστάσεων στην διακυβέρνηση. Θέλουμε να δώσουμε πραγματική κατεύθυνση όσον αφορά τη δημοσιονομική στάση της Ευρωζώνης, ε, τα ενδιαφέροντα, τα ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη και τα οποία ορίζονται από την ετήσια έκθεση. Η Κομισιόν προτείνει τέσσερις συστάσεις για την Ευρωζώνη. Πρώτον, να συνεχιστούν οι πολιτικές που στηρίζουν τη σύγκληση. Δεύτερον, οι, προσα... οι δυνατότητες προσαρμογής και η προσαρμογή των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, καλούμε την εφαρμογή διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές απασχόλησης, στήριξη της απασχόλησης, μείωση του φόρου στα ημερο... στις μισθούς, καθώς και στα αγορές υπηρεσίας για τις δημοσιονομικές πολιτικές θέλουμε να έχουμε ευρύτερα ουδέτερη δημοσιονομική στάση για το 2016 θεωρούμε πως αυτό είναι κατάλληλο για το 2016-2017 να καλέσουμε μείωση στη μείωση του δημοσίου χρέους Τέλος, για τα χρηματοπιστωτικά θέματα, Έχουμε μία σύσταση για μείωση των τοξικών, των μη λειτουργικών δανείων ε, των τραπεζών ε, μέσα στην Ευρωζώνη, ε, καθώς και να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες για την αφαιρεγγιότητα των επιχειρήσεων και οι χώρες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο χρέος να προσπαθήσουν να προχωρήσουν στην εξηγήνση μη βιώσιμων ιδιωτικών τραπεζών. Αυτά είναι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις για σήμερα. Και δίνω το λόγο πίσω στον κύριο Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αμέσως θα δώσω το λόγο στη Μαριάννα Τάισεν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί Πρόεδροι. Αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ξεκινήσω επισημένοντας την οικονομική απόδοση και τις κοινωνικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχει μεγάλη ανισορροπία. Ενώ δηλαδή η απασχόληση και η κοινωνική ασφάλιση σταδιακά βελτιώνονται, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία. Εκεί εξακολουθούμε να έχουμε ανεργία των νέων ε, της του 30% και παραπάνω. Η Σουηδία και η Εστονία τα καταφέρουν αρκετά καλά στο να αντιμετωπίσουν τη μακροχρόνια ανεργία ενώ η Ιταλία και η Φινλανδία δεν έχουν ικανοποιητικά στοιχεία για μακροχρόνια άνεργους. Πρέπει λοιπόν να ανατραπεί αυτή η τάση, να μην διευρύνεται το φάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη, η σύγκληση προς τα πάνω, αυτό χρειαζόμαστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες και ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας στο σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να βαδίζουν χέρι-χέρι. Είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος και γι' αυτό η Κομισιόν είναι ακράδαντα πεπισμένη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αυτού του έτους κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή την κοινωνική δικαιοσύνη την τοποθετεί στο πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης. Και να ε, επισημάνω το εξής στις επενδύσεις. Θέλουμε προτεραιότητα των επενδύσεων χωρίς όμως να ξεχνάμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις συναφείς κοινωνικές επενδύσεις. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να επιταχύνουν, να συνεχίσουν τις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων. Υπολείπονται ακόμα πολλά για την ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια. Η επισφαλής θέσεις απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν θέσει εργασία χωρίς καμία ασφάλεια. Βεβαίως παράλληλα με, την, με τις επισφαλείς θέσεις ε, απασχόλησης υπάρχει και η αδήλωτη εργασία. Ε, είχα ήδη την ευκαιρία να συγχαρώ τον εισηγητή σήμερα το πρωί και το παραλαμβάνω και πάλι εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Για τους μακροχρόνια άνεργους πρέπει να επανέλθουν οι άνθρωποι αυτοί σε δουλειές, είναι προτεραιότητα. Η μακροχρόνια ανεργία είναι το 50% πλέον της ανεργίας και αυτό είναι απαράδεικτο όχι μόνο από ανθρώπινη και κοινωνική σκοπιά, αυτό μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Ε, είμαι αισιόδοξη ότι το Συμβούλιο θα δεχτεί πριν από το τέλος του έτους τις ε, προτάσεις μας όπου αναφέρονται συγκεκριμένα βήματα για να ε, βοηθηθούν οι μακροχρόνια άνεργοι και να επανέλθουν σε θέσεις απασχόλησης. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να διευκολύνουμε τη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας και να καλύψουμε τις κενές θέσεις. Οι διαπραγματεύσεις ε, έχουν μόλις ολοκληρωθεί, οι σχετικές ε, και έχουν ακριβώ αυτό ως στόχο, αυτό που σας είπα. Εξακολουθούμε να έχουμε δύο εκατομμύρια κενές θέσεις παρά τα εκατομμύρια των ανέργων. Αυτό οφείλεται εν μέρη το ότι ε, οι αναζητούντες εργασία δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε ε, στο σχετικό θεματολόγιο που θα συζητηθεί στις αρχές του επόμενου έτους. Επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται ε, στο όριο της φτώχειας. Άρα δηλαδή και εκεί υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωση της ανεργίας την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη βελτίωση των συστημάτων κοινωνικών παροχών. Όσοι λοιπόν είναι μακριά από την αγορά εργασίας πρέπει να τους βοηθήσουμε και αυτούς που έχουν πληγεί από την κρίση και παράλληλα να είμαστε έτοιμοι να αφομοιώσουμε τους πρόσφυγες. Θεωρώ λοιπόν ότι η αποτελεσματική αφομοίωση αυτών είναι καθοριστική σημασίας για θέματα ε, συντάξεων και άλλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες Θέλουμε να είναι βιώσιμη η κοινωνική προστασία, να είναι ικανοποιητική για αυτή τη γενιά και για την επόμενη. Για τα φορολογικά πρέπει ε, η φορολογία ε, να απομακρυνθεί από χαμηλά εισοδήματα και να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Επιπλέον θέλω να υπογραμμίσω ότι ιδιαίτερη σημασία οφείλουμε να αποδώσουμε σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής δικαιοσύνης στις ε, συγκεκριμένες προτάσεις ε, για την Ευρωζώνη. Σημασία αποδίδουμε και στον μηχανισμό έγκυρης προειδοποίησης. Τώρα εξετάζουμε καλύτερα τους κοινωνικούς δείκτες όπως ανεργία των νέων, μακροχρόνια ανεργία, και ποσοστό ε, απασχόλησης ε, στην ανάλυση των μακροοικονομιών ανισορροπιών. Με τον τρόπο αυτό θα κατανοήσουμε καλύτερα και την απασχόληση και τις κοινωνικές επιπτώσεις και προκλήσεις. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά εννοούμε όταν μιλάμε για το να λάβουμε υπόψη μας την κοινωνική διάσταση. Αυτά δεν σημαίνουν μόνο ε, κοινωνικές και νομοθετικές προτάσεις, αλλά σημαίνουν ότι εξετάζουμε τις επιπτώσεις ε, των προτάσεών μας στους ανθρώπους. Σκληρή δουλειά για όλους, για σας, το Κοινοβούλιο, για την Κομισιόν, για τα κράτη-μέλη, για τους κοινωνικούς εταίρους τους οποίους καλούμε να συνεργαστούν μαζί μας. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι οι άνθρωποι να αρχίσουν να αισθάνονται τις προσπάθειές μας στην καθημερινή τους ζωή. Πολύ ωραία. Τώρα, ο εισηγητής ε, της Επιτροπής ΕΚΟΝ, η Μαρία Χουάο Ροντρίγκε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ άλλους καθώς και τον ε, να σας ευχαριστήσω για που ήρθατε και αλλά και τον Μάικλ που έχει συνεργαστεί μαζί μας όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των εκθέσεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και νομίζω πως αυτή η δεύτερη φάση <coughs> συνομιλίας ανάμεσα στην Κομισιόν ε, και το Κοινοβούλιο είναι μια πρακτική η οποία οπωσδήποτε βοηθά σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, υπάρχουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, ναι, αλλά η ανάκαμψη είναι εξαιρετικά περιορισμένη για να μπορέσει να απορροφήσει την ενεργία που έχουμε. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια πιο πράσινη και ευφιέστερη οικονομία όπως λέει και το πρόγραμμα για την Ευρώπη του 2020 αλλά και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. Τώρα, όταν λέτε ότι έχουμε μεγάλα πλεονάσματα στους τρέχοντες λογαριασμούς, ναι, έχουμε επιτυχία στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, αλλά έχουμε και την άλλη του νομίσματος που είναι ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση. Πράγμα το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθούν οι επενδύσει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες αλλά και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θα πρέπει λοιπόν η προσπάθεια να καταβληθεί και από τις δύο πλευρές, και από τις χώρες τις και από τις ελληματικές. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η κατάσταση με μια δημοσιονομική στάση καθώς και μια ομαδοποιημένη οικονομική στάση που βασίζεται στην ε, δημοσιονομική ευθύνη αλλά και που θα προωθεί την υψηλότερη ανάπτυξη, την ισχυρότερη ανάκαμψη αλλά και μια ε, πραγματική ανωδική ε, τάση να ζητήσουμε δηλαδή από τα κράτη-μέλη να να προβούν σε επενδύσεις αλλά και να κάνουν και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα απελευθερώσουν δυναμικό και θα εξασφαλίσουν πιο βιώσιμα ε, συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Όλες αυτές είναι προτάσεις, η νέα όθηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα έπρεπε να εμπλέξουν του Ευρωπαίου πολίτες πολύ πιο άμεσα. Εμείς στο Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι μπορούμε αυτό να το στηρίξουμε και να το προωθήσουμε, αλλά για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα είναι πολύ πιο ε, αναμεμειγμένο όταν πρόκειται για τις συστάσεις αναχώρα αλλά και για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης καθώς και ε, για τις ε, προτεραιότητες της Ευρωζώνης. Τέλος, όπως είδαμε, ζητάμε και μια πραγματικά διοργανική συμφωνία για την οικονομική διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σοφία Ριμπέιρο από την Επιτροπή Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία και κύριοι Επίτροποι. Ξεκινώ τη σύντομη μου αυτή η παρέμβαση σε αυτή τη κοινή ακρόαση ΕΚΟΝ και ΕΜΠΛ ώστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2016 καθώς αυτή η διαδικασία έτσι αποκτά την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση. Και ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάλυση των θεμάτων απασχόληση και των κοινωνικών υποθέσεων για το 2016 θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε ένα πακέτο δίκαιο όσον αφορά τι επενδύσεις, τα κοινωνικά θέματα και τη δημοσιονομική ε, πειθαρχία δεδομένη τη θετική αυτής ε, εξέλιξη που ξεκίνησε με το εξάμεινο ε, παλιότερα. Επίση, δίνεται μεγάλη εστίαση στην κοινωνική πρόνοια η οποία αναφέρεται οριζόντια στις τρεις προτεραιότητε ώστε να υπάρχει σωματική ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική οικονομία και την πραγματική οικονομία που θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Σε σχέση με την ανάπτυξη της νομαλή της οικονομίας ε, μέχρι το 2020 θέλουμε να δούμε κάποιες προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να δώσουμε ε, ιδιαίτερη σημασία στην απασχόληση, ιδιαίτερα στους ε, νέους και στους άνθρωπους μεγάλης διάρκειας αλλά και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τη διεύρυνση και την κάλυψη των προσφύγων καθώς και τους δείκτες ταινίε. Η Κομισιόν προσεγγίζει αυτά τα θέματα πολύ συγκεκριμένα και δίνει λύσεις πολιτικού τύπου πολύ πιο κοντά στου πολίτες, αντίθετα, μάλλον παράλληλα με τις κοινωνικές ε, ε, μεταρρυθμίσεις αλλά και τις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Θεωρούμε επίσης ότι είναι θετικό το να χρησιμοποιηθούν ε, από θέματα ευρωπαϊκά που θα εστιάσουν όχι μόνο στις υποδομές που θα πρέπει να γίνουν βέβαια και αυτές γιατί είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη αλλά επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης συγχαίρω την Κομισιόν γιατί δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο έγγραφο αυτό την ε, εγγύηση μεγαλύτερης εδαφικής και περιφερειακής ολοκλήρωσης έτσι ώστε να τονίσει τη πολύ σημαντική, ε, το σημαντικό ρόλο των ευρωπαϊκών περιφερειών αλλά ανάλογα με το χαρακτήρα της καθεμιάς ε, περιφέρειας. Γενικά έχουμε μέσο και μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης. Θα πρέπει ωστόσο να αγγιηθούμε τη σταθερότητα στους πολίτες μας, ε, αλλά και στις μελλοντικέ γενναίες αυτών. Γι' αυτό και έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το συγκεκριμένη επίλυση των προβλημάτων που τώρα μας ταλανίζουν και τα οποία μόλις σας ανέφερα. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να μας εξηγήσετε πώς προχωράμε στην πρακτική Πώς θα δούμε κατά πόσο άμεσα έχουν απόδοση αυτά τα μέτρα ώστε να εγγυηθούμε την κοινωνική συνοχή λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη πίεση σε σχέση με την ασφάλεια των πολιτών και την αποδοχή, υποδοχή των προσφύγων. Ε, δεύτερον, για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο εξάμεινο θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα δύο επίπεδα εφαρμογής, το ευρωπαίο και το εθνικό, λειτουργούν σωστά. Και έτσι θα ήθελα λοιπόν στις διάφορους τομείς εφαρμογής, εκτέλεσης που είσαι ο καθένας από σας αρμόδιος, θα μου πείτε πώς θα εγγυηθείτε τη ε, διασύνδεση ανάμεσα στο εθνικό πρόγραμμα και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πώς θα ορίσετε τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ειδικά όταν οι εθνικές πολιτικές αποκλίνουν από τις προτεραιότητες που ορίζονται στο εξάμεινο. Σας ευχαριστώ. Έχετε 8 λεπτά όλοι μαζί, κύριε Πίτο. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, ο Αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, για τη γενική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και για τις προτεραιότητες του εξαμήνου δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Έτσι εκτιμούμε και εμείς την κατάσταση. Είναι μια μετροπαθής ανάκαμψη αυτή που βλέπουμε, δεν είναι όμως αρκετά ισχυρή για να επιτρέψει και την ταχεία μείωση της ανεργίας. Οικονομική, οικονομικές μας προτεραιότητες θα πρέπει εκεί να εστιάσουν, στην ενίσχυση της ανάκαμψης. Άρα, επενδύσεις. Και αυτές είναι και οι προτεραιότητες που προτείνουμε στην τη για την ανάπτυξη ενίσχυση των επενδύσεων και σε επίπεδο κρατών μελών. Η Μαριάν επίσης τόνισε ότι δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην σύγκληση και εντό κρατών μελών, προς τα πάνω βέβαια πάντα σύγκληση, και μεταξύ, αλλά και εντός κρατών μελών για την αντιμετώπιση και των περιφερειακών ανισοτήτων. Είναι κάτι που αναφέρθηκε σε αυτό το πλαίσιο. Και βέβαια δίνοντα νωρίτερα στη δημοσιότητα τι συστάσει για τι χώρε τη Ευρωζώνη, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στι κοινέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι χώρε τη Ευρωζώνη και θέλουμε να ενταχθούν, και ε, πιστεύω ότι αυτό θα γίνει πράξη, να ενταχθούν καλύτερα στα εθνικά έγγραφα οι κοινέ αυτέ προκλήσει. Νομίζω δηλαδή ότι ίδια, στο ίδιο μικρό σχήματο κινούμαστε για πολλά από τα ζητήματα. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Ο Πιέρ Μοσκοβισή. Για να ολοκληρώσω, να συμπληρώσω μάλλον αυτά που είπε ο ε, πρέπει να σας πω ότι από το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει συστάσεις για τις χώρες Ευρωζώνης συνολικά. Ο πρόεδρος Γιούγκερ ε, στην πρόσφατη ομιλία για την κατάσταση στην Ένωση υπεσχέθη ότι δεν θα μείνουμε στα λόγια, ούτε θα ε, είναι κενά τα λόγια μας, αλλά θα προτείνουμε συγκεκριμένους προσανατολικούς και κατευθύνσεις να έχουμε μαδοποιημένο προσανατολισμό ε, σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά για την Ευρωζώνη. Το Νοέμβριο δημοσιεύονται τα στοιχεία όπως και τις επισκόπηση για την ανάπτυξη, αναλυφθούν υπόψη εθνικές αλλά και ευρωπαϊκή διάσταση με στόχο ήδη να μπορούμε να έχουμε συστάσεις για την Ευρωζώνη και να συζητηθούν αυτές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και θέλουμε να ενισχύσουμε την επιτυχία αυτή και αυτό θα κάνουμε και στις προτάσεις μας ε, για τη διακυβέρνηση στις χώρες της Ευρωζώνης. Και Τάισεν, σας ευχαριστώ. Τι να προσθέσω τώρα σε όσα ήδη υπόθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό και παραπάνω από συμβολικό ότι μιλάμε για ανάκαψη και σύγκληση στον τίτλο και της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη, είναι σημαντικό και να το πούμε αυτό. Και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ε, στο πακέτο συνολικά. Έχουμε λοιπόν ένα νέο στοιχείο τη σύγκληση. Ήδη είχαμε προσπαθήσει και κατά το παρελθόν να εργαστούμε με στόχο τη σύγκληση και είχαμε μερικώ επιτύχει. Είχαμε την πολιτική συνοχή στα διαδροτικά ταμεία και πριν την κρίση είδαμε ότι υπήρχε μια προσέγγιση μεταξύ των κρατών Λόγω τη κρίση όμω πάλι απομακρύνθηκαν τα κράτη-μέλη και βλέπουμε και αύξηση των ανισορροπιών και ανισοτήτων και μέσα στην ίδια χώρα. Αυτό δεν είναι καλό για την κοινωνία και τη συνοχή, ούτε για την ανάπτυξη είναι καλό. Πάρα πολύ ανισορροπία και ανισότητα φρενάρει την ε, ανάπτυξη. Το έχουν πει πολλοί θεσμοί, πολλοί φορεί και εκεί θα εστιάσουμε σιγά σιγά θα προχωρήσουμε, θα δούμε ποιοι είναι οι δείκτες, ε, και τα κριτήρια, τα benchmarks που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βέβαια όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όπως και τις επιδόσεις των κρατών μελών. Τώρα σε ό,τι αφορά την κοινωνική ε, προστασία και ασφάλιση νομίζω ότι δίνουμε έμφαση στον τομέα αυτό και στις ε, εκθέσεις αναχώρα εστιάζουμε και στη βιωσιμότητα και τη διάρκεια των συστημάτων. Θέλουμε να δούμε βιώσιμα ασφαλιστικά συστήματα για το μέλλον, αλλά να δούμε υπάρχει επαρκή σκάλυψη, είναι αρκετά υψηλά τα επιδόματα, είναι αποτελεσματικό το σύστημα, εξυπηρετεί τους στόχους που έχουμε ορίσει. Πιστεύω ότι τα κάνουμε όλα αυτά και αυτό καταδεικνύει ότι λαμβάνουμε υπόψη και το κοινωνικό σκέλος. Επίσης τονίζουμε και την καταπολέμηση της ανεργίας, Έχουμε τη μακροχρόνια ανεργία και την ανεργία των νέων. Είναι δύο πολύ σημαντικά προβλήματα και μας έχουν απασχολήσει και εξακολουθούν να μας απασχολούν και το εξάμεινο και η επισκόπηση για την ανάπτυξη. Επίσης, επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο μεταξύ άλλων. Φυσικά το λαμβάνουμε αυτό υπόψη και ρητά το αναφέρουμε και στο έγγραφο που εγκρίναμε την προηγούμενη Πέμπτη. Αν δείτε δε τους στρατηγικούς τομείς στους οποίους ε, μπορούμε να επενδύσουμε, αναφέρεται εδώ. Το πακέτο για τις επενδύσεις, μάλλον το Ταμείο Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, που ξεκίνησε φέτος, νομίζω ότι και αυτό προσφέρει εχέγγυα για επενδύσεις ε, σε ανθρώπινο κεφάλαιο, άρα πρέπει να πω ότι ε, λογικά θα πρέπει να καθησυχάζονται με αυτόν τον τρόπο οι ανησυχίες των εισηγητών. Ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Τώρα οι ερωτώντες έχουν 1,5 λεπτό στη διάθεσή τους, αυστηρά. Ο κύριος Χαφιέ Λόπες είναι ο πρώτος ερωτών. Ο Σέργιο Κουτιέρης δεν μπορούσε να είναι εδώ. Θα πω εγώ κάποια σχόλια ε, σχετικά με όσα είπατε και με τις εκθέσεις που μας παρουσιάσετε. Πρώτα απ' όλα ε, συμφωνούμε και μας ε, είπατε ότι είναι προτεραιότητα κοινωνική δικαιοσύνη και η σύγκληση προς τα πάνω και τα κοινωνικά πρότυπα. Συμφωνούμε αυτές τις προτεραιότητες. Το θέμα είναι πώς αυτό θα γίνει πράξη. Κοινωνική προστασία ε, με μακροοικονομικές πολύ σαφές προϋποθέσεις που τις συζητούμε, πώς αυτά θα τα συνδυάσουμε και πώς θα έχουμε αυτή τη σύγκληση προς τα πάνω και πώς θα προχωρήσουμε με συγκεκριμένα προγράμματα όπως το Mobility Package για παράδειγμα δεν τα εκτελούμε αυτά τα προγράμματα παρότι πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεύτερο, γνωρίζουμε ότι η ανάκτηση πράγματι είναι ευθραυστή, είναι ε, βραδία, υπάρχουν εποχικοί παράγοντες και από τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που ζητούνται με βάση την ασφάλεια και την ευελιξία ε, συμφωνούμε ε, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια σε αυτό τον πίνακα όμως υπάρχουν προβλήματα επισφάλειας, έχουμε προσωρινές ε, συμβάσεις ε, ορισμένου χρόνου, έχουμε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Οι διαρθωτικές λοιπόν μεταρρυθμίσεις πώς ε, από τη θεωρία θα περάσουν στην πράξη. Και έχουμε ένα πρόβλημα, επαναλαμβάνουμε, την επισφαλή εργασία, γιατί περί τέτοια εργασία μιλάμε. Και έχουμε και ασθενή ανά, ανάκαμψη, επαναλαμβάνω. Επίσης, μας εξηγήσατε ποιο είναι ένα από τα προβλήματα και ανισορροπίες που υπάρχουν έχουμε το πλεόνασμα στους τρεχούμενους λογαριασμούς και μία από τις λύσεις που προτείνεται είναι η κατανάλωση, επενδύσεις, πώς μπορούμε να τονώσουμε δηλαδή ε, κατανάλωση και επενδύσεις σε κάποιες χώρες. Το ερώτημα όμως, ε, σε κάποιες ε, περιπτώσεις, γιατί επιμένουμε, εδώ γιατί δεν επιμένουμε για να αυξηθούν οι μισθοί παραδείγματο χάρη που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε και εκμεταλλεύτηκε τις έρευνες προηγούμενων ετών. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή επιβεβαιώνει τις προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί για εφέτος δηλαδή επενδύσεις, ε, δημοσιονομική σταθεροποίηση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή απόφαση να δοθεί σημασία σε αυτές τις ε, προτεραιότητες. Και έχω μια ερώτηση που αφορά ε, σε αυτές τις τρεις σημαντικές προτεραιότητες. Πρώτον, εάν εστιάσουμε στις επενδύσεις, γνωρίζετε ότι οι επενδύσεις ε, στον ιδιωτικό τομέα ήταν φιδωλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην Ευρωζώνη. Και γι' αυτό λοιπόν ρωτώ, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να επενδύσει περισσότερο, να ξεπεραστεί αυτή η επιφυλακτικότητα. Ενώ ε, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτίθεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη αφορά στην οικειοποίηση, εθνική ιδιοκτησία αν θέλετε των ε, μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι οι συστάσεις αναχώρα χώρα δεν εφαρμόζονται σωστά. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει έτσι ώστε να προσφέρει κίνητρα στα κρατη για να συμμετέχουν και αυτά περισσότερο στην εφαρμογή ε, των ε, αναχώρα συστάσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε για την Ευρωζώνη, αυτή τη στιγμή ε, έχουμε ένα ικανοποιητικό κλίμα και πρέπει κανείς να αντιρωτηθεί τότε ε, γιατί παρόλα αυτά ε, ορισμένες χώρες δεν τα καταφέρνουν καλά. Η Ελλάδα, ας πούμε, είναι οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Στη Γαλλία αυξάνεται η ανεργία, ε, σε σχέση με τους ε, προηγούμενους ε, μήνες έχει αυξηθεί κατά πολύ. Κρύγνονται τα χρέη στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες από τότε που ο Γαλλίας ανέλαβε το αξίωμά του αυξήθηκε το δημόσιο χρέος της Γαλλίας κατά 250 δισεκατομμύρια. Ούτε και στους άνεργους βλέπουμε καμιά βελτίωση. Οι νέοι εγκαταλείπουν τις ε, χώρες αυτές και πηγαίνουν εκεί που έχουν κάποια ελπίδα. Κατανοώ βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάπως να κρατήσει τα ενία, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι λόγω του υψηλού χρέους, ε, της αδυναμίας για μεταρρυθμίσεις, ε, δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Δύο ερωτήσεις. Η μία προς τον κύριο Μοσκοβισή. Μετά από 8 χρόνια η Γαλλία ε, που δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τα κριτήρια λόγω της, ε, του προσφυγικού, της προσφυγικής κρίσης προτίθεται να αναστείλει το σύστημα. Ε, αυτό αν γίνει τελικά δεν θα ισχύει κανένας κανόνας περιχρέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ποιοι είναι οι στόχοι σας για να μπορέσετε να επανέλθετε στην πεπατημένη. Και η δεύτερη ερώτησή μου στους δύο άλλους επιτρόπους. Όλο και περισσότερο καταβάλλονται προσπάθειες αυτή η αδυναμία για μεταρρυθμίσεις να αρθεί κυρίως ε, μέσα από την αμοιβεοποίηση των κοινωνικών συστημάτων. Και πώς λοιπόν μπορείτε να διατηρήσετε την ανταγωνιστικότητα, την ευελιξία και την αρχή της επικουρικότητας. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Σήμερα έχουμε να κάνουμε με την ετήσια έκθεση ανάπτυξης του 16. Τη διάβασα την έκθεση και εκεί ε, υπάρχουν πολλά που μοιάζουν να είναι συμπαθητικά. Βέβαια, ε, μου θύμισε αυτή η έκθεση το πενταετές της ε, Ντεντέρ του 51 γιατί εκεί γίνεται λόγος για χάρτη πορείας, ε, για πρωτοβουλίες, για σχέδια με εθνικά στοιχεία, για πλατφόρμες, για μέτρα πρόθεση και ανταλλαγής μεθόδων. Γίνεται λόγος για νέες τεχνολογίες, για την αηφορία και αυτό που δεν εκπλήσει γίνεται και παραπομπή σε άλλες εκθέσει. Άρα δηλαδή λίγα λόγια, στην έκθεση αυτή γίνεται λόγος για καθορισμό συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και η έκθεση χρησιμοποιεί ε, αυτή την ορολογία που χρησιμοποιούσαν οι παλιές ε, κεντρικά κατευθυνόμενες οικονομίες. Εγώ νομίζω ότι πάει τέλειος αυτό με την ε, αλλαγή των καθεστώτων. Εγώ τάσομαι υπέρ του να υπάρχει μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς γιατί μόνο αν μια οικονομία είναι ελεύθερη από κεντρικά κατευθυνόμενο προγραμματισμό, μόνο έτσι θα υπάρχει κοινωνική και οικονομική ελευθερία. Εσείς τι θέλετε, το θέλετε κι εσείς αυτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντομπρόσκης. Uh, okay. Uh, number of uh, questions Αρκετές ερωτήσεις ε, εστιάζουν στην οικονομία. Καταρχήν πώς θα επιτύχουμε την σύγκληση προς τα πάνω. Έχουμε δύο ομάδες που εργάζονται σε αυτό. Η μία ασχολείται με το πώς θα χρησιμοποιήσει καλύτερα τους δείκτες ε, στην μακροοικονομική μας διαδικασία και μακροοικονομική μας ανάλυση, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές και πτυχές και πτυχές της απασχόλησης ε, καλύτερα και το άλλο με τη, ε, την μεγαλύτερη χρήση του benchmarking, ε, της ε, σύγκρισης επιδόσεων, να δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι καλύτεροι μαθητές, αλλά και πώς το κατάφεραν έτσι ώστε το benchmarking να είναι πιο πολύ δεσμευτικό νομικά. Και τέλος η ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης. Επίσης βάζουμε στους ε, λογαριασμούς των κρατών μελών περισσότερους πόρους ώστε να αντιμετωπίσουν ε, τα τις κοινωνικές ή τις περιφερειακές ανισορροπίες. Βλέπουμε δηλαδή από κοινού ε, τις οικονομικές και τις κοινωνικές πτυχές των θεμάτων. Θεωρούμε πως αυτά τα δύο συνδέονται, είναι αλληλένδετα τι μέτρα λαμβάνουμε ώστε να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα. Σε πολλές χώρες έχουμε διαφορετικές προκλήσεις. Σε κάθε χώρα μάλλον έχουμε διαφορετικές επενδυτικές προκλήσεις και γι' αυτό τώρα προετοιμάζουμε μια έκθεση για τις προκλήσεις της επενδυτικές στα διάφορα μέλη ώστε στη συνέχεια να εξετάσουμε με ποιους τρόπους θα τις αντιμετωπίσουμε. Ίσως όμως να μην είναι ένα θέμα το οποίο να είναι το ίδιο σε όλα τα κατημέλη, είναι πιο ειδικό για κάθε κράτος και γι' αυτό και κάνουμε ατομικές μεμονωμένες εκθέσεις για να εξετάσουμε ανά περίπτωση την κατάσταση. Για την εφαρμογή των CSR στον αναχώρα συστάσεων, ναι, αυτή είναι μια κλασική ερώτηση. σημαίνει βασικά καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε χώρα και εφαρμογή των κατάλληλων ε, μέτρων και συστάσεων. Τώρα, για τις προτεραιότητες για τις προτεραιότητες των εξαμήνων και τις ε, λύσεις θα έλεγα πως ε, Ε, θα έλεγα πως ε, η επισκόπηση για την ανάπτυξη αποτελεί μια βάση για το πώς λειτουργεί η ε, Ευρώπη, οι χώρες μας, ο κ. Μασκοβησή. Ναι, τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την μακροοικονομική ανισορροπία. Θεωρούμε ότι τα πλονίσματα τρέχοντας του συζυγίου είναι κάτι το χαρακτηριστικό και δεν επιτρέπει ισορροπημένη ανάπτυξη. Γι' αυτό και το λόγο μάλιστα σκεφτόμαστε μέτρα τα οποία επιτρέπουν τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης, δηλαδή επενδύσεις, ε, κατάρτιση ε, και ό,τι επίσης ενθαρρύνει τις επενδύσεις ευρύτερα. Όσον αφορά τις επενδύσεις, να θυμίσω το πόσο επίκαιρο και σωστό είναι το σχέδιο Juncker και ο συνδυασμός ιδιωτικών με δημόσιες επενδύσεις επενδύσεις. Έχουμε ήδη ε, χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο πρότυπο. Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες. Ε, οι ιδιωτικέ όσο γίνεται περισσότερο ε, και οι δημόσιε μόνο εκεί που είναι απολύτω απαραίτητο. Έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη απόδειση. Τώρα όσον αφορά τις αναχώρα συστάσεις. Η φιλοσοφία μας είναι να τις απλοποιήσουμε, να τις καταστήσουμε πιο στρατηγικής φύσης, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Έπειτα άκουσα τόσο είπατε για τη Γαλλία. Ε, εγώ νομίζω πω θα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μα και τη λογική μα. Στη Γαλλία επίση πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσει, αλλά η Γαλλία είναι και η δεύτερη οικονομία τη Ευρωζώνης. Είναι μια χώρα που γνωρίζει ανάκαμψη όπω κι άλλε, αν και ε, θα επιθυμούσαμε ίσω να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική η οικονομική τη πολιτική, θα πρέπει να γίνουν και εκεί ε, μεταρρυθμίσει. Και δεν άκουσα να γίνεται λόγο από πλευρά του Προέδρου τη Δημοκρατία για οποιαδήποτε ε, άλλη λύση. Άκουσα από εκείνον ότι η ασφάλεια, γιατί μια χώρα όταν ε, πλήττεται από τέτοιες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις καθιστά την ασφάλεια πρωταρχική της προτεραιότητας. Νομίζω πως η αξιοπρέπεια και η πια ο ανθρωπισμός απαιτούν να τα ακούσουμε αυτό και να μην ψάχνουμε να βρούμε έτη και το τέλος του Συμφώνου Σταθερότητας πίσω από όλα αυτά που υπόθηκαν είναι η κυρία Τάισεν. Σας ευχαριστώ. Να, να συμπληρώσω αυτά που υπόθηκαν. Ζητείτε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και λέτε, λαμβάνω υπόψη αυτήν την παράμετρο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά για την Ελλάδα Έχουμε μπροστά μας μια νέα συμφωνία με την Ελλάδα για να μιλά της που Δεσμεύτηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρξουν και άλλα προγράμματα να γίνει μελέτη αντικτύπου για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το γεγονός ότι έχουμε τρεις δείκτες κοινωνικούς από το scoreboard λοιπόν σε σαφείς δείκτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, γιατί θα μπορέσουμε έτσι να αξιολογήσουμε και την κοινωνική διάσταση στα κράτη-μέλη και να λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα. Οι κοινωνικοί συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και αυτό δείχνει ότι τους λαμβάνουμε υπόψη, λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις τους σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό για να μπορέσουμε να βρούμε τις σωστές ισορροπίες. Ο συνάδελφος Λόπεθ για την αύξηση των μισθών σε κάποιες χώρες. Ναι, φυσικά και πρέπει να γίνει αυτό. Δεν έχουμε όμως εμείς αρμοδιότητα, δεν είναι ευρωπαϊκή αυτή αρμοδιότητα όπως ξέρετε, είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα αυτό. Σε ό,τι αφορά τι ανισορροπίε, γίνεται σαφή διάκριση μεταξύ κρατών μελών που έχουν πλεόνασμα, κρατών μελών που έχουν ε, έλλειμμα. Και προτείνουμε όσοι έχουν πλεόνασμα να μην αποταμιεύουν αλλά να επενδύσουν πραγματική οικονομία κατά το δυνατόν. Είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να ε, υπάρχουν ομοιόμορφα κοινωνικά μοντέλα. Όχι, δεν το είπαμε αυτό, δεν θα το διαβάσετε πουθενά. Εμείς είπαμε απλά ότι πρέπει να έρθουν πιο κοντά οι χώρες, ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ανισορροπίες και οι ανισότητες. Δεν είπαμε ότι θέλουμε ομοιόμορφα ε, σχήματα και συστήματα, γιατί ο στόχος μας δεν είναι η αρμόνιση, αλλά η σύγκληση. Τα, κράτη, τα, μελη είναι κύριοι ε, του τρόπου και των μέσων που χρησιμοποιούν. Εμείς επαναλαμβάνω βλέπουμε αν υπάρχει επαρκής κάλυψη, αν υπάρχουν προβλήματα και αν αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν και άλλα κράτη-μέλη και αν αυτό ισχύει σίγουρα πρέπει να δοθεί δέουσα προσοχή, επενδυτικό κλίμα. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να πω ότι φυσικά και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Οι αποφάσεις για τις επενδύσεις είναι πολύ πρέπει να πληρούνται ορισμένε προϋποθέσεις. Νομίζω ότι στην Ευρώπη πρέπει να μπορούμε και εμείς ε, να επηρεάζουμε τα πράγματα και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Η Ένωση Κεφαλαιογορών, Ψηφιακή Ένωση, Ενεργειακή Ένωση, Κυκλική Οικονομία, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ε, πολιτική απασχόληση και ανάπτυξη. Ε, δίνουν κίνητρα για προσλήψεις και θα πρέπει σίγουρα και οι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν να έχουν και τι κατάλληλε δεξιότητε. και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκτήσουν αυτέ τι δεξιότητε. Και εδώ μιλάμε και για καινοτομία μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Μαρία Χάρκιν, 1,5 λεπτό, αλλά εκπροσωπείτε και τη δική σα πολιτική ομάδα για τα ζητήματα τη ΕΚΟΝ και τη κλιματική αλλαγή. άρα θα σα δώσω τρία λεπτά συνολικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιτρόπους που ήρθαν σήμερα εδώ και για τις εξηγήσει που μας έδωσαν. Ε, θέλω να σας πω, με χαρά μου διαβάζω, ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στα θέματα απασχόλησης και κοινωνικής φύσεως. Η κυρία Τάισεν μίλησε για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη που πρέπει να συμβαδίζουν. Ε, Διαβάζοντας λοιπόν ε, τις εκθέσεις που έχουν κυκλοφορήσει, αυτό είναι το οδηγό νήμα που τις διατρέχει. Έτσι λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ε, στην κοινή έκθεση για την απασχόληση αναφέρεται ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο να εξυγχρονίσουν την αγορά εργασίας, αλλά δεν αντιμετωπίζουν συστηματικά τις ανισότητες ε, ε, δεν καταλαβαίνω όμω τι ακριβώ είναι οι ανισότητε και μετά γίνεται λόγο για insider και outsider. Πώ ε, προτίθεστε να το αλλάξετε αυτό. Δεν λέω ότι αυτό έχετε κατά νου, αλλά περίπου ένα χρόνο νωρίτερα εδώ μία νέα κοπέλα από την Πορτογαλία μίλησε γι' αυτό και είπε μήπω ε, εννοούν ότι ε, θα απολύσουν τους γονείς μας για να βρούμε εμεί δουλειά. Δεν λέω ότι αυτό έχετε κατά νου, αλλά θα ήθελα λιγάκι να μας το εξηγήσετε αυτό. Και επίση τι είδου μέτρα μπορούν να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες. Δεύτερον, όσον αφορά τις επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Και πάλι διαβάζω την κοινή ε, έκθεση για την απασχόληση και εκεί αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια η ε, απασχόληση αφορούσε ε, συμβάσεις εργασίας και όχι μόνιμες θέσεις απασχόλησης και λέει ε, ότι αργότε, η έκθεση της, μάλλον η αύξηση της απασχόλησης αφορά κυρίως την αύξηση των συμβάσεων εργασίας, συμβάσεις έργου. Εκεί υπήρξε αύξηση από το 16% περίπου στο 19%. Πάντως τα στοιχεία σοκάρουν τα γενικά στοιχεία. Και ε, στο πλαίσιο και της πρώτης μου ερώτησης για τους insider και τους outsider στην αγορά εργασίας θα ήθελα να γνωρίζω τελικά τι προτείνει η Κομισιόν για να αντιμετωπιστούν ε, αυτά τα στοιχεία που σοκάρουν. Η άλλη μου ερώτηση έχει σχέση με το θέμα των πλεονασμάτων στην Ευρωζώνη. Ε, ακούσαμε ότι υπάρχει ε, πλεόνασμα του ισοζυγίου τραχουσών σε είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Μας είπαν επίσης ε, ότι πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητε και να στηριχτεί η ανάκαμψη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνο ε, παρατεταμένη ε, περιορισμένης ανάπτυξης. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό θα μειωθεί από χώρε οι οποίε μπορούν να αυξήσουν τις επενδύσεις και τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν από αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαντιμούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μοσχοβησή, η Κομισιόν παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες την πρόταση για μια, ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Και λίγες ώρες μετά αυτή η πρόταση της Κομισιόν διάχθηκε μια πολύ επιθετική κριτική με πλήρη άρνηση από τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σόιμπλε. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτή την σπουδή του κ. Σόιμπλε να επιτεθεί και να αρνηθεί την πρόταση της Κομισιόν. Σκοπεύετε να επιμείνετε στην πρότασή σας, που αποτελεί και μια δέσμευσή σας, ή θα κάνετε πίσω, επειδή σας μάλωσε ο κ. Σόιμπλε. Για την κυρία Τίσεν, πριν από λίγο καιρό ο Ιταλός Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Παντοάν, κατέθεσε μια πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα στήριξης των ανέργων που να λειτουργεί συνδυαστικά με τις προσπάθειες των κρατών μελών έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η αυξημένη ανεργία. Πώς βλέπετε ως αρμόδια επίτροπος την πρόταση Παντοάν, θα την εξετάσει η Κομισιόν, τη βλέπετε θετικά. Και η τρίτη μου ερώτηση πάλι προς τον κύριο Μοσκοβισή. Γύρω από τα θέματα του χρέους, η Κομισιόν θεωρεί ότι το χρέος δυσκολεύει την ανάκαμψη επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις που χρειάζονται. Είναι διατεθειμένη η Κομισιόν στην περίπτωση της Ελλάδας να παίξει έναν μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ζητά μια γενναία ελάφρυση του ελληνικού χρέους και το Eurogroup που αρνείται μια τέτοια ιδέα. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Έλληνας, είπε ότι το Φεβρουάριο μπορούμε σε αυτά τα θέματα να έχουμε μια παραγωγική συζήτηση. Θα εργαστείτε γι' αυτό. Thank you. I'll give the floor to Madam Zimmer. The floor is yours. Yeah, Ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος Τάισεν επισήμανε προηγουμένως ότι τα κράτη-μέλη φέρνουν την ευθύνη για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά το μεταξύ έχουμε προχωρήσει. Από το 2010 και εντεύθεν έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν κοινοί δείκτες, ότι υπάρχουν κριτήρια, ότι υπάρχει μια στρατηγική για την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά από όλα αυτά δεν βλέπουμε τίποτα να υπάρχει σε αυτή την ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ονοματίζεται το ε, την κοινωνική ανάπτυξη, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σύγκληση και κάτι άλλο. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι επανέρχεται μία θέση, μία άποψη, η περίφημη flex security, η ευελιξία με ασφάλεια. Δεν χρησιμοποιείται αυτόν τον όρο, αλλά ακριβώ αυτό περιγράφεται. Τα τελευταία χρόνια η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια δεν βοήθησε στο να διασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης και ούτε οι εργαζόμενοι ένιωσαν τέτοια ασφάλεια έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε μια διαδικασία καινοτομιών. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο σε τελική ανάλυση γιατί μιλάτε συνεχώς για ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί δεν μιλάτε για δημόσιες και κοινωνικές επενδύσεις, γιατί δεν προβάλλετε αυτά τα δύο είδη επενδύσεων, γιατί ε, κάθε δημόσια επένδυση αποφέρει 1,2 μέχρι 1,3 επιπρόσθετη ανάπτυξη. Όταν υπάρχουν δημόσιες αυξάνονται και ιδιωτικές επενδύσεις. Μήπως στους δείκτες θα έπρεπε να υπάρχει κι άλλος ένας δείκτης που να αφορά τις δημόσιες επενδύσεις και κάτι άλλο. Έχω, έχω άλλο ένα ερώτημα. Ισχύει το ότι το πακέτο κινητικότητας, το mobility package ε, θα παραταθεί ή μάλλον ούτε καν θα ληφθεί υπόψη ε, ίσως γιατί αυτό έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη και την σύγκληση ανάμεσα στην οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη. Ο Επίτροπος και Αντιπρόεδρος κύριος ε, Ντομπρόφσκης. Για το θέμα το πλεονάσματο της Ευρωζώνης και του κατά πόσο αυτό έχει ε, αντίκτυπο και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα αυτό δεν είναι νέο στο θεματολογιό μας, ε, αν δούμε και τις φετινές αναχώρα συστάσεις, ε, αλλά και αυτές των προηγούμενων ετών, οι πλανασματικές χώρες ε, δέχονται συστάσεις ώστε να σταματήσουν τις δημόσιες επενδύσεις και να κινητοποιήσουν την επιτυχή της ζήτησης της οικονομίας τους. Σαφώ σε μια οικονομία πρέπει να εξετάζουμε όλες τις πλευρέ και να προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Αυτό αναφέρεται και στην ε, ετήσια επισκόπηση. Τώρα, για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων και τις επικρίσεις που δέχεται. Όταν προετοιμάζαμε αυτή την πρόταση, εξετάζαμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις ανησυχίες ε, όσον αφορά τον κίνδυνο των, ε, για τις χώρες που δεν είχαν ε, τηρήσει τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα εθνικά τους προγράμματα και νομίζω πως είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην έκθεσή μας αρκετά δηλαδή από αυτά τα στοιχεία τα αντιμετωπίζουμε λέγοντας ότι αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων θα είναι προσβάσιμο προσιτό μόνο στις τράπεζες από τα κράτη-μέλη που έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους υπό την Τραπεζική Ένωση, δηλαδή αν έχουν εθνικό πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων, δηλαδή μεταγραφή του BRT, ε, BRT της οδηγίας BRD, με συγχωρείτε, και επίσης ε, ε, αυτές οι τράπεζες ε, συμβάλλουν περισσότερο στο σύστημα κοινής, στο κοινό σύστημα ασφάλισης ή συνασφάλισης. Τώρα, επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες είναι η προτεραιότητά μας και προσπαθούμε να τις παροτρύνουμε και τις δύο. Η συμβουλή μας είναι να δοθεί προτεραιότητα στις δαπάνες που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη και οι δημόσιες επενδύσεις φυσικά είναι τμήμα αυτών των δαπανών που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη. Επίτροπος Στάισεν, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όσον αφορά την αγορά εργασία, την πρώτη ερώτηση της κυρίας Χόκκιν. Αυτή η αγορά εργασία με τους insider και τους outsider, πράγματι τη χρησιμοποίησαμε αυτή την ορολογία, γιατί υπάρχει πόλωση στην αγορά εργασία, διότι οι νέες συμβάσεις είναι επισφαλείς, είναι μερικής απασχόλησης. Οι άνθρωποι μετακινούνται από μία σύμβαση έργου στην επόμενη και δεν έχουν μέλλον. Ε, δεν έχουν προοπτική ούτε για σταθερή θέση απασχόλησης ούτε για καλύτερο μισθό. Επίσης δεν έχουν προοπτικές για περαιτέρω κατάρτιση για να μπορούν να οργανώσουν καλύτερα την ε, ζωή τους. Υπάρχει λοιπόν μια ανισορροπία που ενισχύεται συνεχώς. Ε, αυτό ισχύει στα κρατημέλη και γι' αυτό ε, πρέπει όλοι να μεριμνήσουν έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα σύστημα αυτών που είναι μέσα και αυτών που είναι έξω, των ins και των out, ε, δηλαδή κάποιοι να την χάνουν απόλυτης προστασίας και άλλοι καθόλου προστασίας. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό, εκείνο το οποίο κατά παρελθόν ορίζαμε ως άτυπες μορφές απασχόλησης, θα το ορίζουμε ως και τυπικές ε, θέσεις απασχόλησης. Πολλοί θα λένε, συγγνώμη, αυτές οι συμβάσεις έργου δεν είναι και τόσο κακές, ε, γιατί αν με αυτές ε, προκύπτει ανάπτυξη, γιατί όχι. Αν όμως οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να αποκτήσουν καλύτερη θέση απασχόλησης, αν δηλαδή αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου βλά υπάρχει εκμετάλλευση, ε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε έτσι ώστε να επικρατεί ισορροπία και θα πρέπει να μεριμνήσουμε για το κατά πόσον οι νόμοι που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανοποιητικοί για να στηρίξουν τις θέσεις μας. Ο τελικός στόχος είναι τελικά ε, να υπάρχει ισορροπία, ε, να υπάρχει σταθερότητα, ασφάλεια, flex security, αναφέρθηκε αυτό και γνωρίζουμε ότι η αγορά εργασίας είναι σημαντική, βεβαίως και αλλάζει η κοινωνία, βεβαίως και αλλάζει και η αγορά εργασίας, όλα αλλάζουν. Και γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να είμαστε ευπροσάρμοστοι. Αυτό ισχύει όπως σας είπα και στην αγορά εργασίας. Με πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης να είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι όταν θα χρειάζονται υποστήριξη, όταν θα χρειάζονται κοινωνική προστασία, να υπάρχει αυτή η κοινωνική προστασία. Αυτό εμείς κατανοούμε με την ευελιξία και την ασφάλεια. Κατά τα άλλα, όσον αφορά αυτά τα δύο θέματα, βεβαίως και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους κοινωνικού εταίρους, αυτοί καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και ε, τέθηκε ένα ερώτημα τι θα γίνει τελικά με την πρόταση, θα την αναδιατυπώσω, δεν την πω ακριβώς όπως ελέγχθη, με την πρόταση ένα τμήμα της ε, ανεργίας να αμοιβεοποιηθεί με την έννοια ότι να τον αλάβουν ε, όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή αμοιβεοποίηση του επιδόματος εργασίας. Υπάρχει μια τέτοια ε, πρόταση να υπάρχει ένα ειδικό ταμείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα χρησιμοποιείται για έκτακτες καταστάσεις, για σοκ. Τώρα, κατά πόσον από εκεί θα μπορούν να εκταμιεύονται επιδόματα ανεργία. Ξέρετε, αυτό δεν συζητήθηκε ακόμα τόσο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σας λέω, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σύγκληση ε, όσον αφορά Τη ε, ενέργεια των κρατών μελών πριν καταλήξουμε και εμεί σε μια συγκεκριμένη πρόταση. Ο κύριο Μοσκοβισή. Δύο απαντήσεις, πολύ γρήγορα για την εγγύηση των καταθέσεων καταρχάς. Όταν δρομολογήσαμε την Τραπεζική Ένωση ήταν τρει οι πυλώνε τη, ήταν σαφέ αυτό. Ό,τι αφορά την εποπτεία, εξυγίανση που σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, θέλουμε την ε, Bridge Finance να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ήταν ε, εγγύηση καταθέσεων. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση ε, που είναι φιλόδοξη και σοβαρή. Ο Wolfgang Schäuble έκανε τις παρατηρήσεις του, για το θέμα αυτό. Σίγουρα θα ξεκινήσει η συζήτηση και για τους δύο πλώνες δεν ήταν εύκολα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και οι συνάδελφοί μου είναι πάρα πολλοί πραγματιστές. Τώρα σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρέος. Έχουμε ένα χρόνο διάγραμμα, έχουμε προθεσμίες και η λογική είναι ότι πρώτα πρέπει να πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις και να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Ήδη λοιπόν είχαμε μια πρώτη δέσμη μέτρων που ψηφίστηκε δεύτερη δέσμη μέτρων ε, αυτή τη στιγμή θα ε, βρίσκεται στην διαδικασία έγκρισης. Πολύ, στεν, ε, πολύ φιλόδοξες και πολύ θαραλές μεταρρυθμίσεις και για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και πιστεύουμε ότι είναι προς την καλή κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να έχουμε σημαντικές εκταμιεύσεις ε, για την εφαρμογή του προγράμματος και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και μετά θα δούμε και το ζήτημα του χρέους και εύχομαι και ελπίζω να γίνει το συντομότερο δυνατό και νομίζω ότι στις αρχές του έτους θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Για να πώ θα ολοκληρώσουμε τώρα τη συζήτηση δεν το ξέρουμε, ακόμα θα το δούμε. Tyson again on the Για το πακέτο κινητικότητας. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για το πακέτο κινητικότητα ξέχασα να απαντήσω. Να σας ε, διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι. Είχαμε μια συζήτηση προσανατολισμού στην Επιτροπή και συμφωνήσαμε ότι θα προτείνουμε ένα πακέτο. Αυτή είναι η θέση τη ε, Κομισιόν. Θα γίνει αυτό, θα κατατεθεί ένα πακέτο ε, που θα αφορά την πληροφόρηση, την αναθεώρηση στόχων για την οδηγία απόσπασης εργαζομένων, αναθεώρηση ε, της οδηγίας για το συντονισμό ε, στην κοινωνική ασφάλιση κτλ. Θα ήμασταν έτοιμοι μέσα στο μήνα, αλλά όπως ξέρετε υπήρξαν απρόβλεπτα ζητήματα, ασφάλεια, ε, πρόσφυγες, είναι πολλά τα ζητήματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό και δεν έχει μπει ακόμη στην ημερήσια διάταξη επόμενη εβδομάδα στο θέμα από ό,τι γνωρίζω. Είμαστε όμω έτοιμοι και από τη στιγμή ε, που θα το ε, έχουμε καταρτήσει θα το παρουσιάσουμε στο Κοινοβούλιο. Ε, okay. then we proceed to... Να περάσουμε στην Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους επιτρόπους για την παρουσία της. Σήμερα ακούσαμε ότι ε, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, που είναι σημαντικός και οι εξελίξεις ε, είναι γνωστές. Θα θυμάστε όμως ότι πέρυσι είχαμε πάρει την υπόσχεση ότι θα υπάρξουν κατευθυντήρες γραμμές για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών γιατί μιλάμε για τον κοινωνικό τομέα, δεν είναι μόνο η απασχόληση. Τι έγινε με αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ για την κοινωνία των πολιτών, τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Επίση, σε σχέση και με αυτό που είπε η συνάδελφο Γκάμπι Τσίμερ, τα θέματα που αφορούν τη φτώχεια. Οι επίτροποι θεωρούν ότι η ανάλυση των προτινόμενων αλλαγών ε, των πολιτικών των κρατών μελών έχουν εξεταστεί υπό το πρίσμα του πώς επηρεάζουν τα επίπεδα της φτώχειας. Απλά να γίνεται μια αναφορά, δεν θέλουμε μάλλον να γίνεται απλά μια αναφορά, αλλά έχει γίνει και μια ανάλυση. Επίση, ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ οικονομική και κοινωνικού σκέλου. Εγώ θέλω να προσθέσω και την περιβαλλοντική διάσταση, ίσω να μην σα εκπλήσει αυτό. Αρχίζουν ε, στην COP21 οι σημαντικέ συζητήσει. Ε, αύριο δημοσιεύεται το πακέτο για την κυκλική οικονομία. Το ανέφερε και Τάισεν. Διαρωτώ με, αν λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά μηνύματα που μπορούμε να δώσουμε για τη διεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε, για τις δεξιότητες, τις θέσεις εργασίας, ε, το τα κτλ. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι όλα αυτά ότι ε, στην επισκόπηση της ανάπτυξης και στη διαδικασία του εξαμήνου και αν όχι, τι υποτίθεται να κάνετε για να αλλάξει την κατάσταση. Φίλιπ Λάμπερτς τώρα. Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω αγγλικά θα μιλήσω με, για την κακιά λέξη που αρχίζει από χ, χρέος, που δεν μειώνεται από το 2009 και μετά το λένε και τα έγγραφά σας. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι σημάδι επιτυχία του πολιτικού μείγματο ε, που έχετε εφαρμόσει ε, εδώ και κάποια χρόνια. Ε, το σκέφτεστε καθόλου, σας απασχολεί ή απλά καλύψετε την ίδια κατεύθυνση. Και επειδή έχω χρόνο για μια δεύτερη δυσάρεστη ερώτηση, θα μιλήσω για το πλεόνασμα. Είπατε ναι, ναι, μα ανησυχούν τα πλεονάσματα τη Γερμανία και άλλων χωρών που αυξάνονται κατακόρυφα. Ο κ. Μοσκοβισή έλεγε ότι δεν οδηγεί σε ισορροπημένη ανάπτυξη. Τι θα πει αυτό δεν ξέρω, αλλά τέλο πάντων λέτε ότι σα ανησυχεί το θέμα αυτό. Τι κάνει η Γερμανία με την ανησυχία σα, Μάλλον όχι και πολλά. Γιατί εξακολουθεί να αυξάνεται κατακόρυφα το πλεόνασμα τη Γερμανία. Σα ανησυχεί μεν, αλλά τι θα κάνετε δε. Απλά θα παρακολουθείτε ως θεατές αυτά που γίνονται. Ευχαριστώ. I give the floor to... Ε, Να δώσω τώρα το λόγο στον Ντομινίκ Μαρτά. Ευχαριστώ. Κάνετε μια τυπο αντικειμενική διαπίστωση που είναι πάντα ίδια, δεν επαρκούν οι επενδύσει, ενθυμική είναι η ανεργία, σημαντικέ μακροοικονομικέ ανισορροπίε και μα φέρνετε λίγο πολύ τι ίδιε λύσει σε οικονομική σύγκληση, φορολογική σύγκληση, κοινωνική σύγκληση. Και μα μιλάτε όλο και ε, περισσότερο για την κρίση του 2008 και συνέχεια το ίδιο αναφέρεται σαν να έχει ε, περάσει να ήταν μια κακή στιγμή, μια συγκυριακή κρίση κάνετε λάθος. Δεν είναι καθόλου συγκυριακή αυτή η κρίση, είναι δομική, είναι διαρθρωτική κρίση, ακριβώς λόγω αυτών των συγκλήσεων που δεν πετυχαίνεται μεταξύ των κρατών μελών, οικονομική, φορολογική, δημοσιονομική και κοινωνική σύγκληση. Αντίθετα λοιπόν έχουμε τώρα μία συγκυριακή κρίση, η κυρία Τάισεν πρέπει να το ξέρει αυτό, και είναι η προσφυγική κρίση. Συγκεκριμένα λοιπόν, τι θα κάνετε για να απορροφηθούν αυτοί οι πρόσφυγες χωρίς να διευρυνθούν ακόμη περισσότερο οι ανισορροπίες για τις οποίες εκφράζετε την λύπη σας. Πολύ ικανοποιημένοι είμαστε που μας είπατε ότι πέφτουν τα μέσα δημοσιονομικά ελλείμματα και φτάνουν στο 1,7% του ΑΕΠ. Ο κύριος Μοσκοβίση απάντησε πριν, θα επιμείνω όμως, λυπάμαι γιατί δεν με ικανοποίησε, ήταν σαφής απάντησή σας. Ο πρόεδρος Ολάντα πολύ ξεκάθαρα είπε ότι πρέπει το σύμφωνο ασφάλειας να προηγηθείτε του συμφώνου σταθερότητας. Δεν ήσασταν πολύ ξεκάθαρο στην δική σας απάντηση. Πώς πιστεύετε και τι θα, ε, μάλλον πώς προτίθεστε να ε, συνοδεύσετε κατά κάποιο τρόπο ε, να υιοθετήσετε αυτά που λέει ο πρόεδρος Ολόντ. Ο μου Μοσκοβής να απαντήσει. Ναι. Για πολλά από τα ερωτήματα Mm. είναι σημαντικά. Το πρώτο αφορούσε το τρέχον πλεόνασμα και μάλιστα το συγκεκριμένο τρέχον πλεόνασμα της Γερμανίας. Δείχνει μία ε, θεαματική ανωδική ε, προεκβολή 7 ή 8% τα δύο τελευταία χρόνια και πιθανότατα γύρω στο 9% για φέτος. Αλλά δεν τίθεται καν ε, θέμα να κατηγορήσουμε την γερμανική οικονομία για την πιο σημαντική λόγω του μεγέθους της και η πιο ανταγωνιστική της υπήρου μας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρίσκεται τελείω παράδοξο να ζητήσουμε από την γερμανική οικονομία να εγκαταλείψει την ανταγωνιστικότητά τη. Αντιθέτω, μπορούμε να διαπιστώσουμε και το κάναμε και πέρσι ότι στην πτυχή τη εσωτερική συζήτηση η γερμανική οικονομία βρισκόταν κάτω από το δυναμικό τη κάτω από τη δυνατότητα της και σας θυμίζω ότι μιλήσαμε πέρσι για τις επενδύσεις, για τις υποδομές, για την κατάρτιση. Έχουμε διαδικασίες στο πλαίσιο της ε, ΜΥΠ που κάναμε εκεί και σημαντική πρόοδο και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Βέβαια, με βάση το αποτέλεσμα. Είναι η αρχή μιας διαδικασίας και όχι το τέλος της. Κανείς δεν ανέφερε αυτή την κρίση ως κυριακή κρίση. Διαρκεί από τα τέλη του 2007. Είναι βιώσιμη, ε, μακρά διαρκείας. Ωστόσο, είπαμε ότι είμαστε στην τρίτη, ε, ε, τρίτη χρονιά, διαδοχική χρονιά θετικής ανάπτυξης και φαίνεται να βελτιώνονται τα πράγματα σε σημαντικό βαθμό. Ωστόσο, θέλουμε περισσότερα και πιο γρήγορα στην Ευρωζώνη. Προφανώς, Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πολιτικών που από τη μια πλευρά επέτρεψαν την ε, σωστή χρηματοδότηση, από την άλλη τη μείωση του ε, ελλείμματος. Και όλα αυτά βεβαίως θα συμπληρώνουμε, όπως ξέρετε, με το σχέδιο Juncker. Με ρωτήσατε ε, τι, κάνει, τι είπε ο Γάλλος πρόεδρος που μίλησε στο Γαλλική Βουλή που όπως ξέρετε ε, ε, έγινε τρεις μέρες μετά από τις αναδιφόρες, τις δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις που κόστησε τη ζωή σε 130 ανθρώπους. Ε, δεν αναφέρθηκε στο σύμφωνο σταθερότητα. Είπε και απλώς ότι έπρεπε μέσα σε αυτό το δραματικό πλαίσιο να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες υπέρ της ασφάλειας στη Γαλλία και ανακοίνωσε μέτρα συγκεκριμένα ο Γαλλός Πρόεδρος τα οποία εγκρίθηκαν από το σύνολο των εθνικών αντιπροσωπιών που το χαιρέτησε ε, και από το σύνολο του Κοινοβουλίου που τον χαιρέτησε όρθιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα αντέδρασε και είπε ότι εφόσον υπήρχαν αυτές οι συνθήκες που ήταν εξαιρετικές, δραματικές και τραγικές, φυσικά και έπρεπε να τις λάβουμε υπόψη με εξαιρετικό και εκτακτό τρόπο. Και αυτό δεν είναι καθόλου αντιφατικό με το Σύμφωνο Σταθερότητας, διότι εάν δείτε αυτά τα 600 εκατομμύρια είναι 0,015 του ΑΕΠ. Και ο Μισελ Σαπά, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, είπε πως η γαλλική πορεία δεν θα επηρεαστεί από αυτό ούτε το 2016 ούτε το 2017. Τη στιγμή που διακυβεύεται η εθνική ενότηση, η αξιοπρέπεια, ε, δεν θέλουμε εδώ να κάνουμε πίσω ούτε να χαλαρώσουμε τα μέτρα για τη Γαλλία. Θέλουμε όμω να βοηθήσουμε τη Γαλλία να ενισχύσει την, ασφάλειά τη. και το σύμφωνο σταθερότητα δεν είναι ένα αυτόσκοπό. Ε, απλά δείχνουμε ότι είμαστε ευφυεί και ανθρώπινοι και όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό νομίζω γιατί έχουμε να κερδίσουμε από, αυτό. Τώρα, όταν σας παρουσιάσαμε τις μακροοικονομικές μας ε, προβλέψεις, ε, δεν είχαμε προβλέψει τους ε, πρόσφυγες. Τότε, πρόκειται για δημόσιες δαπάνες και είναι ένα ε, μια απέτηση για την οικονομία με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθούν πιο ευφυείς πολιτικές ώστε να ενταχθούν αυτοί όλοι οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας, να υπάρξει περισσότερη κατάρτιση και εδώ θα πρέπει να δούμε μια σοβαρή προσέγγιση γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, να συζητήσουμε με τις τρίτες χώρες όπως το κάναμε με την Τουρκία αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι που ήταν απαραίτητο για να περιοριστούν οι ροές αλλά και για να έχουμε μια προσέγγιση που να είναι ε, ε, προσέγγιση ε, υποδοχή για αυτού του ανθρώπου που φεύγουν από ένα καθεστώ που είναι ντροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και που απειλεί τι ζωέ του. Ευχαριστώ. Επίτροπο Επίτροπος Τάισεν. Η Επίτροπος Τάισεν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ σύντομα να απαντήσω σε την, την ερώτηση του κ. Τζιν Λάμπερτ ε, σχετικά με τη φτώχεια, κατά πόσον δηλαδή ε, βλέπουμε τη φτώχεια, κατά πόσον λαμβάνουμε υπόψη μας τις ε, επιπτώσεις στην φτώχεια. Η αντιμετώπιση της φτώχειας είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία εξακολουθεί να καθορίζει την πολιτική μας και αυτό το βλέπει κανείς και στο έγγραφό μας για το πρώτο εξάμεινο του 2016. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες προσπάθειές μας για τη μετώπιση της φτώχειας. Η κρίση βέβαια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Περισσότερες θέσεις απασχόλησης και αποτελεσματικότερα συστήματα προστασίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ε, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής 2020. Ε, Εν τω μεταξύ ε, θα υπάρξει ενδιάμεση αξιολόγηση. Είπαμε ότι δεν θα ξεχάσουμε τους στόχους μας, ακόμα και αν υπήρξαν υπαναχωρήσεις λόγω της κρίσης. Πρέπει όμως να είμαστε φιλόδοξοι. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις, να στηριχθούν τα κράτη-μέλη και να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Όσον αφορά το θέμα των προσφύγων. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο συνάδελφος Μοσχοβησή. Πρέπει να εντάξουμε τους ανθρώπους που έχουν δικαίωμα σε προστασία, διεθνή προστασία, πρέπει να τους ε, εντάξουμε και να τους αφομοιώσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αγορές εργασίες μας και έτσι να μπορέσουν να συμβάλλουν όσο γίνεται πιο σύντομα στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να θέσουμε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 να δημιουργήσουμε τις ε, προϋποθέσεις ώστε να εκείνοι να καταβάλουν την προσπάθεια να μάθουν τη γλώσσα και τα λοιπά, αλλά σημαίνει και από δική μας πλευράς ότι πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να θέλουμε να τους υποδεχτούμε και να τους δώσουμε την πρόσβαση στην αγορά εργασία μας. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί τα κρατημέλη πρέπει να λάβουν αποφάσεις ναι μεν, αλλά υπάρχουν κρατημέλη που θέλουν να περιορίσουν το χρόνο στον οποίο έχουν δικαίωμα οι πρόσφυγες να διζητήσουν ε, διεθνή προστασία προστασία πριν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία. Και υπάρχουν χώρε μέλη που ήδη έχουν σύντομη προθεσμία, ενώ άλλε που έχουν κάνει τέτοιε προτάσει στα κοινοβούλια του. Πιστεύω πως ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε αν θέλουμε να έχουμε συνοχή και να βρούμε και πάλι μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντιπρόεδρος Δομπρόφσκης. Σας ευχαριστώ. Έχουν λεφτεί πάρα πολλά. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα του χρέους. Ήδη φέτος ε, το δημόσιο χρέο στην Ευρώπη κατά μέσο όρο έχει αρχίσει να μειώνεται. Έχουμε δει για αρκετά χρόνια συνέχεια να μειώνεται το έλλειμμα. Για του χρόνου υπολογίζεται ότι θα φτάσει στο 1,7 του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος ε, αναμένεται να περιοριστεί. Τώρα, επειδή ε, οι χώρες γίνονται έτσι πιο ευάλωτες σε ε, ένα νέο οικονομικό σοκ. Θα πρέπει να πούμε ότι το 60% του χρέους Μάλλον, το χρέος μπορεί να είναι στο 60% του ΑΕΠ. Τώρα όμως στην Ένωση φτάνουμε και στο 90% του, ψηλού, του χρέους, γι' αυτό πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να το μειώσουμε στις, στις χώρες που έχουν πρόβλημα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντανούτα για Σλοβιέσκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιτρόπους για την παρουσία τους. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και συμφωνώ απόλυτα με την Επίτροπο Τάισεν για το ανθρώπινο κεφάλαιο που είναι και το μεγαλύτερο δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αποτελέσει θεμέλιο μιας ε, ισχυρής ανταγωνιστικής Ευρώπης. Έχουν τεθεί τα ερωτήματα που θέλω να θέσω λίγο, κάπου, λίγο διαφορετικά σε ό,τι αφορά το flex security, την ευελιξία με ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Φυσικά οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και η ασφάλεια είναι παράγοντες ε, αναγκαίοι για τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την Ευρώπη και να τις ε, απαγορεύσουμε να υιοθετήσει ευέλικτες μορφές απασχόλησης γιατί πρόκειται για μια διεθνή τάση. Όμως αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας θα πρέπει να είναι ασφαλείς, ιδίω για την ασφαλόθεση θέση εργασία. εργασίας. Επίσης, νομίζω ότι πιο πολλά θα πρέπει να μιλάμε για την ε, ασφαλή ευέλικτη και όχι την ευέλικτη ασφάλεια. Και να λάβουμε υπόψη μα και τα δημογραφικά προβλήματα. Ξεργάζεστε κάποιε συστάσει, είπατε, ε, αναχώρα. Βλέπετε και τι γίνεται στο παγκόσμιο προσκήνιο. Υπάρχουν καλά παραδείγματα ασφαλούς ε, και ευέλικτης απασχόλησης από άλλες χώρες του κόσμου. Μια άλλη ερώτηση τώρα που απευθύνω σε όλους τους επιτρόπους. Ε, αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος μία μείζωνα κρίση την μεταναστευτική. Αυτό τι είναι, ευκαιρία ή απειλή για την Ευρώπη. Θα πρέπει να χαραχθεί μία πολιτική ένταξης, ολοκλήρωσης, ε, ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασία. Έχουμε εμπειρίες άλλες καλές, άλλες κακές. Ε, πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε, να τις αξιοποιήσουμε το συστάτω το θέμα αυτό με τι χώρε μέσα στο πλαίσιο των συστάσεων χώρα γιατί πολλέ φορέ οι βέλτιστες πρακτικέ δεν διαδίδονται από τη μια χώρα στην άλλη και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι ζωέ μεταναστών θα έχουν πολύ σημαντικέ επιπτώσει στην οικονομική μα κατάσταση και στου προπολογισμού. Η Μπάρμπαρα Πάπελ, ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροπη με την Μητής Επισκόπηση για την Ανάπτυξη βλέπετε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τον οικονομικό προσανατολισμό, δημοσιονομική εξυγίανεση, επενδύσεις. Αν δούμε όμως τις προοπτικές που δημοσίευσε το φθινόπωρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι τόσο ρόδινες. Ελάχιστη είναι η ανάπτυξη. Από το 1,9 φτάνει το 1,6. Μειώνεται η ε, ελεύθερη πτώση των τιμών των πρώτων υλών, ε, η πτώση της τιμής του ευρώ ένα του δολαρίου, ε, ανεργία παρόλα αυτά μεγάλη σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, ε, Ελλάδα, ούτε και η Γαλλία ούτε, και αυτή πληρεί όλα τα κριτήρια, άρα πόρο απέχει σύγκληση, 18 χώρες έχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, δύο παραπάνω από πέρυσι, παρά τα δισεκατομμύρια επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και παρά τα μέτρα συντονισμού ρύθμισης ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και ε, Ανάπτυξης ε, απέδειξα ε, ότι είχε λόγο ύπαρξης, ε, έχει φέρει αποτελέσματα. Τι έχετε να μας ε, προτείνετε για μεγαλύτερη σύγκληση και για ανάκαμψη. Θα κύριος Φέρμπερ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Είπατε είναι προτεραιότητες, βελτίωση του πνευματικού κλίματος, διαθετικές μεταρρυθμίσεις και το φορολογικό φορολογικό στην φορολογική βελτίωση. Δεν είμαι προφήτη, αλλά θα τολμήσω να κάνω μια ε, πρόβλεψη για του χρόνου. θα έχουμε ακριβώ τα ίδια προβλήματα και το θέμα ε, με την διαδικασία αυτή ε, είναι όταν διαπιστώνουμε ότι τελικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος, δεν εφαρμόζονται συστάσεις αναχώρα, δεν εφαρμόζονται οι στόχοι για τον προπολογισμό μακροχρόνιες επενδύσεις ε, και στο ιδιωτικό ε, τομέα ε, πάλι καθυστερούμε, πολύ αργή πρόοδος. Τι θα κάνει συγκεκριμένα η Κομισιόν τους επόμενους μήνες για να υπάρξει το πατούμενο πλαίσιο του χρόνου να έχουμε άλλες και χτισίες προτεραιότητες. Thank you. And the last question, uh, or... Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Η κοινή έκθεση καθώς και η έκθεση για τον μηχανισμό προειδοποίησης που περιλαμβάνει και νέους και ειρωνικούς δείκτες δείχνει βελτιώσεις ε, όσον αφορά την ανεργία και δείχνει επίσης πως υπάρχει σαφής συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα αποτελέσματα και την εφαρμογή της εγγύησης για τους νέους και της πρωτοβουλία για τους νέους, ε, για την απασχόληση των νέων στα κρατημέλη. Είναι σαφές ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική και ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Τα κρατημέλη χρειάζεται διαρκώ να του υπενθυμίζουμε τις ε, δεσμεύσεις του σε αυτό το μέτωπο, αλλά και να τα στηρίξουμε οικονομικά για να αντιμετωπίσουν πολιτικά το θέμα αυτό. Να σας ρωτήσω λοιπόν ακριβώς για αυτό το θέμα, Επίτροπε Τάισεν. Θεωρείτε με αυτέ τι προοπτικέ και αυτή την κατάσταση, την, την εισήγηση νέων περαιτέρω στοχευμένων μέτρων, εκτό από αυτά που ήδη έχουν ε, να εγκριθεί για την προχρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων ώστε να διευκολυνθούν τα κράτη να εφαρμόσουν καλύτερα την εγγύηση για τους νέους και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων όσον αφορά κυρίως την ποιότητα της εφαρμογής. Ευχαριστώ. Θα αρχίσουμε με τον Επίτροπο Μοσχοβησή. Από τον τελευταίο γύρο. <coughs> Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη γιατί θα χρειαστεί να σας αφήσω. Να απαντήσω να σας ε, μιλήσω για την κατάσταση της διαδικασίας ε, που αναφέρθηκε από τον κύριο Φέρμπερ. Μπορεί να μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Σίγουρα πρέπει να απλοποιήσουμε, να είμαστε πιο στρατηγικοί και επίσης να πείσουμε, να βελτιώσουμε το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο. Ο, ο Βάλτης θα σας πει τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν, αλλά ίσως να είμαι λιγότερο αρνητικός ε, για τα αποτελέσματά μας. Όταν διαπιστώνω και συγκρίνω τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καταρχήν δημόσια οικονομία σε σχέση με αυτό που έγινε τις προηγούμενες χρονιές, διαπιστώνω πως ο αριθμός των κρατών για, που είναι σε έλλειμμα μειώνεται. Και το έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό του, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, τώρα είναι πολύ πιο κάτω από το 3% και μένουν μόνο τρεις χώρες που είναι πάνω από αυτό το όριο. Επίσης διαπιστώνουμε πως για πρώτη φορά το επίπεδο του δημόσιου χρέους αρχίζει να μειώνεται και η αντιστροφή θα τονιστεί ακόμη περισσότερο στο 2017. Η ανάπτυξη αρχίζει να αναπτερώνεται με ένα ρυθμό του 2% που δεν είναι αρκετό, αλλά πάντως είναι αρκετά σταθερό. Και αυτό καθοδηγήθηκε από εσωτερικού ανέμους, διαπιστώνουμε ακόμα ότι αρχίζει να κάμπτεται και η ανεργία Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι οι στρατηγικές μας δεν είναι πανάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν βοηθήσει να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρέπει ακόμα περισσότερο να προσπαθούν και αυτό είναι ε, το στόχο της διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματο, αλλά και της ε, ε, διαδικασίας του εξαμήνου. Σα ευχαριστώ κυρία. Κύριε Τάισεν, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω στην κυρία Βαλιοβεύσκα ότι κάθε μέρα εξετάζουμε την κατάσταση στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά την ανεργία πάνω απ' όλα εστιάζουμε στα δεδομένα της γενικής ανεργίας. Αλλά υπάρχουν και δικοί στόχοι για την αντιμετώπιση τη μακροχρόνια ανδρία και τη ανδρία των νέων. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση νομίζω, χρησιμοποιούμε και τα διαρθρωτικά ταμεία, ταμεία δηλαδή ιδίω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ξέρουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν απαντήσεις στις ειδικές τάσεις αναχώρα. Πρέπει να στηρίξουμε τι καλε πρακτικέ και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν στο σωστό δρόμο. Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, τον κύριο Μποναφέ, είμαστε στο τέλη του 2015. Η εγγύηση για την νεολαία δεσμεύτηκαν να λάβουν για αυτήν δομικά μέτρα τα κρατη μέσα σε κάποιους μήνες. Θα διατυπώσουν προτάσεις για να βοηθήσουν τους νέους που κάνουν τη μετάβαση από το σχολείο και το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας. Για την ανεργία των νέων έχουμε δείκτες, ίσως περισσότερες από όσους χρειάζονται, για να δούμε κατά πόσον έχουμε επιτύχει ή όχι τους επιδιωκόμενους στόχους, αν έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε προεξοφλήσει. Συλλέγουμε τα στοιχεία και το 16 θα γίνει έκθεση αφού συλλέξουμε τα δεδομένα από τα κράτη-μέλη. Θέλουμε οι πολιτικές μας να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, σε πραγματικά και αντικειμενικά δεδομένα. Τα συλλέγουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία τώρα, μετά θα, ε, θα υποβάλουμε την έκθεσή μας στο κοινοβούλιο και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε την πολιτική αυτή ή μήπως χρειαστεί να αλλάξουμε ε, τακτική και έχουμε και την ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου όπως γνωρίζετε Έχουμε ήδη δώσει ε, κονδύλια για την πρωτοβουλία για τους νέους ε, των προτέρων και θα δούμε αν χρειάζονται κονδύλια και το 2016. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η δουλειά αυτή. Κύριος Ντομπρόφσκης. Okay. Ε, ε, thank you very much. So first the... Κοιτάξτε, όσον αφορά την μακροοικονομική πολιτική και τις σχετικές προτεραιότητες, βασιζόμαστε στις ε, προτεραιότητες ε, του περασμένου και αυτού του έτους. Γιατί πιστεύουμε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εξακολουθούν να είναι ίδιες, δηλαδή εξακολουθούμε να έχουμε μια συγκρατημένη ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς είναι δυνατόν να ενισχύσουμε αυτήν την ανάπτυξη. Μετά, για θέματα που έχουν σχέση με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Εδώ υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες ε, που παίζουν ε, θετικό ρόλο, χαμηλά επιτόκια, χαμηλές τιμές πετρελαίου, ε, χαμηλή ισοτιμία του ευρώ, καλά αυτά, αλλά βέβαια υπάρχουν και αρνητικές εξελίξεις, υπάρχει η επιβράντηση ανάπτυξης των αντιόμενων οικονομιών, η αστάθεια στην ε, περιοχή μας όσον αφορά τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αλλά αστάθεια και όσον αφορά τις ε, γείτονές μας προς Ανατολάς. Αναφέρομαι στην ε, διένεξη Ρωσίας-Ουκρανίας. Όλα αυτά επηρεάζουν την οικονομική μας ανάπτυξη και τις σχετικές προβλέψεις. Όσον αφορά τώρα στο να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάθος ανάλυση σε 18 κράτη-μέλη, δηλαδή σε δύο περισσότερα από ό,τι κατά ε, τα προηγούμενα έτη, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι γίνεται σε βάθος ε, ανάλυση, αυτό δεν ε, προδιαγράφει το αποτέλεσμα. Επίσης, αυτό δεν σημαίνει ότι μια χώρα μπορεί ε, χωρίς περαιτέρω λόγο να βγει από αυτή την αυστηρή επιτήρηση. Είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε το κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών για το 2016. Σε γενικές πάντως γραμμές πρέπει να πω ότι οι προτεραιότητες τη ευρωπαϊκή Επιτροπής να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να επαναφέρει τη διαδικασία της σύγκλησης, οι προσπάθειες αυτές μοιάζουν να την χάνουν υποστήριξης και από τις Επιτροπές Έκων και Απασχόλησης. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και για να προχωρήσουμε τις πολιτικές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς και εμείς που παρακολουθήσατε αυτή την κοινή επιτροπή θα επανέλθουμε όταν ε, ε, θα έχουν τεθεί νέα ερωτήματα και ίσως και με αποτελέσματα, γιατί φλεγόμαστε γι' αυτά. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας στο Κοινοβούλιο και είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα κάνετε και στην Επιτροπή. Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε αποτελέσματα το συντομότερο γιατί ένας είναι ο στόχος ο στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, η οποία συνδέεται στενά με αυτό που είναι ο βασικός μας στόχος στην Ένωση, δηλαδή η δημοκρατία. Δεν μπορούμε να ε, κάνουμε τίποτα με την ανεργία αν υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν σήμερα εδώ και θα τα ξαναπούμε σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα όλων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.